Κύριε Κυρία Πρόεδρε των Ίσων Μάρσαλ, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπουργέ Ντάλι, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Συμφωνία του Παρισιού είναι ένα ιστορικό επίτευγμα της διεθνούς κοινότητας. Η πρώτη στην ιστορία παγκόσμια δέσμευση